Il Presidente. Care colleghe, cari colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ξεκινάει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιδημία ισχυρή και ακόλη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Επίτροπο Ντάλι για πέντε λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις